εβδομάδα στην ατζέντα και το έχουμε βάλει χωστό σήμερα. Πρόκειται για την ε, ε, επίσκεψη της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ασία και τη σχετική έκθεση, η οποία έχει κατευθεί εδώ ως έκθεση για την επίσκεψη των Παγκλαντές. Να πούμε όμως ότι πήγαμε και δύο ημέρες στις Μαλδίβες, όπου θα ήθελα να υποδείξω στους συναδέλφους ότι το ένα μέρος που επισκεφθήκαμε πέρα από τη συνάντηση με τους ε, πολιτικούς της ΜΚΟ και τα μέλη της ε, κοινωνίας των πολιτών ήταν μια φυλακή. Για να διευκρινίσω ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης της Μαλδίβες στον Μπαγκλαντές. Να πω ότι έγιναν υψηλόβαθμες συναντήσεις και με την Πρωθυπουργό την ίδια και με τον Υπουργό Εξωτερικών Εμπορίο και θα ξέρετε ότι έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα ναι. και την πρόεδρο του Κοινοβουλίου και με την, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία, λέει ο πρόεδρος. Συναντηθήκαμε με εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών, θα σας πω κι άλλα γι' αυτό, με τον επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος του Μπαγκλατές και έγιναν και συναντήσεις με εκπρόσωπους του τομέα της κλωστοφαντουργίας και του τομέα της ε, κατασκευής έτοιμων ενδυμάτων και επίσης επισκεφτήκαμε και βρισοδεψία στην ΤΑΚΑ και διάφορα project τα οποία επιδοτούνται από τον ΟΗΕ και έγινε και μία συνέντευξη τύπου στο τέλος της επίσκεψης και η οποία και περιλάμβανε 62 στοιχεία σε ανακοίνωση τύπου. Πολύ μεγάλη διαφορά με το τι συμβαίνει συνήθως στις Βρυξέλλες. Συζητήσαμε προφανώς θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κοινωνία των πολιτών ήταν πολύ πιο απρόθυμη να σαντηθεί μαζί μας σε σχέση με το παρελθόν και αυτό πρέπει να το αποδώσουμε σε μία μείωση του δημόσιου χώρου. Θέσαμε θέματα περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης σε ό,τι αφορά και τελοφωνίες κάποιων bloggers. Ζητήσαμε να μας διευκρινίσουν την ποιότητα των ερευνών. Θέσαμε θέματα για την ενδεχόμενη άνοδο του εξτρεμισμού. Πρόκειται για μια χώρα όπου υπάρχει μεγάλη ανεκτικότητα και που σκοπός είναι να αυξηθεί για παράδειγμα ο βουδιστικός τουρισμός. Θέσαμε το θέμα της επιβολής της αντικής ε, ποινής, το είχαμε θέσει και στο παρελθόν με την Πρωθυπουργό και πώς μπορεί να γίνει μια συζήτηση τουλάχιστον στη χώρα σε ό,τι αφορά το εμπόριο, το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλήσαμε και για το μέλλον της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων το οποίο και αποτελεί ε, έναν εξάρτητο σώμα το οποίο απολαμβάνει υψηλού κύρους στο Μπαγκλαντές και τονίσαμε την ανάγκη να υπάρχουν ανεξάρτητοι θεσμοί σε ό,τι αφορά και θέματα της εκλογικής επιτροπής. Θα ξέρετε ενδεχομένως ότι δεν χρηματοδοτείται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση το σώμα αυτό λόγω ανησυχιών. Θέσαμε το θέμα της πολιτικής κατάστασης όπου πολλοί έχουν την αίσθηση ότι τα περιστατικά βίας του τελευταίου έτους μετά τις εκλογές προκάλεσαν μια μετατόπιση σημαντική στην χώρα σε ό,τι αφορά τον τομέα της κατασκευής και παραγωγής ενδυμάτων μιλήσαμε για τους όρους ε, βιωσιμότητα στους οποίου καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελούν τα συντηρητικά μέσα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρουμε ότι έγιναν πολλές επιθεωρήσεις και εφαρμόστηκαν πολλά προγράμματα διόρθωση, αλλά πολλέ πολλές χρειάζονται ακόμα. Η παραγωγή όμως τονίζουν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία μετά το 2018. Επίσης, πήραμε μαζί μας και την, τον κύριο Καρύμ που είναι επικεφαλής των θεμάτων εμπορίου για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα και σε ό,τι αφορά το ενεχόμενο καθεστώς GSP+, ένα σύστημα κινητευμένων προτιμήσεων ε, με κάποια επιπρόσθετα στοιχεία και προνόμια. Θέσαμε το θέμα της διαφθοράς μεταξύ άλλων, αλλά είδαμε και την εξέλιξη ενός ε, ε, επιχειρηματικού συμβουλίου με τις ΗΠΑ, στο οποίο παρακολουθούμε πάρα πολύ. Η Ινδία, Μιανμάρ, η κατάσταση Ραχίνγκα, δεδομένου ότι το Μπαγκλατές ε, έχει υποδεχθεί από τη Βερμανία 300.000 και πλέον πρόσφυγες. Και νομίζω ότι αυτά είναι επιγραμματικά τα ζητήματα. Προφανώς και θέσαμε και άλλα ζητήματα, αλλά ξέρω ότι περιμένουν οι συνάδελφοι να ξεκινήσει η ψηφοφορία και ότι υποτίθεται ότι θα γινόταν πριν από κάποια λεπτά. Έχει ξεκινήσει ήδη η ψηφοφορία αυτή. Θα σταματήσω λοιπόν και είμαι φυσικά στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σακοράφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ε, θέλω να επισημάνω ένα πρόβλημα που έχω εντοπίσει και, ε, και έχει δημιουργηθεί φυσικά όσον αφορά στην ακρίβεια και την αξιοπιστία, αν θέλετε, της μετάφρασης της έκθεσης προόδου και κατ' επέκταση και των τροπολογιών που ακολουθούν την έκθεση από την Αγγλική στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, γλώσσε. Για αυτό το θέμα έχω ήδη κάνει ε, επιστολή στου αρμόδιου φορεί και στις αρμόδιε υπηρεσίες. Η τροπολογία 114 που έχω καταθέσει στα ελληνικά δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια στην αγγλική γλώσσα. Έχει παραποιηθεί η τροπολογία που έχω καταθέσει κύριε Πρόεδρε, ε, πουθενά εγώ προσωπικά δεν αναφέρω τη φράση «Μακεδονική δημόσια διοίκηση» και θα παρακαλούσα την γραμματεία να επιληφθεί πάρα αυτά του θέματος, διότι για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Κύριε Βάγγελ, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω απλώς εσάς ως Πρόεδρο και τους συναδέλφους της Επιτροπής για την απόφαση που έγινε προηγουμένως να αναβληθεί η ψηφοφορία για αυτή την έκθεση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ξέρετε, υπήρξε μια κομβική χρονική στιγμή όταν το Κοινοβούλιο της Μακεδονίας αποφάσισε να αναβάλει τις εκλογές, τις πρόορες εκλογές εκεί και θέσπισε μια νέα ημερομηνία για τις 5 Ιουνίου του έτους αυτού. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο διότι ήταν κοινή η αξιολόγηση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προετοιμασίες για την εκλογική διαδικασία δεν είχαν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε οι εκλογές θα μπορούσαν να τηρήσουν τα υψηλά επίπεδα δημοκρατίας, διαφάνειας και κράτους δικαίου. Έχουμε τώρα μια νέα ημερομηνία, 6 Ιουνίου διορθώνει ο μιλτής, όχι 5 Ιουνίου. Και έχω καταθέσει δύο προφορικές τροπολογίες που αναφέρονται σε αυτή την αλλαγή ημερομηνία και επίση αναφέρονται στην παρατήρησή μα ότι ήταν απαραίτητο η διαδικασία αυτή ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία προσέγγιση τη Μακεδονία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν όλα τα κόμματα στη χώρα αυτή. Και οι προφορικέ ερωτήσει βρίσκονται στον κατάλογο ψηφοφοριών. Περαιτέρω παρατηρήσεις, όχι, ας ψηφίσουμε. Να περάσουμε στην τροπολογία 13. Χάουιτ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65. 64 θέλετε έλεγχο για την 64. Έλεγχο ηλεκτρονικό για την 64. I think ότι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ποτέ όμως δεν αρκούν οι ψήφοι από το ΕΛΚ. Αστείευεται ο Πρόεδρος. Οκ. Okay. Μάλιστα. 64. Εγκρίνεται με διαφορά. 66. 66. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 με προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 79 λοιπόν τώρα. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρασε εγκρίνεται 30 υπέρ 21 κατά. Συμβιβαστική 5 με προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 τώρα. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 32 κατά απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Δεν έχω 112 ο πρόεδρος. Α, μάλιστα. Η Κόβατσεφ. 112 υπέρ. Στον κατάλογο του ΕΛΚ έχουμε ένα πρόβλημα νομίζω αλλά εν πάση είναι 112. Κόβατσεφ. 112. Ε, Υπέρ. Μα ψηφίστε τουλάχιστον εσείς κύριε Κόβατσεφ. Τελευταία ευκαιρία. Υπερψηφίστε εσείς τουλάχιστον. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορία. 24 υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. Κύριε Κόβατσεφ, αν δεν είχατε διστάσει θα είχατε κερδίσει. 113. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 114. Υπέρ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ.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 Κατά. Άποχες έγκρινεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 138. Υπέρ. Κάτα. Άποχες. Έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen πέρα ψηφοφορία. εγκρίνεται με 34 υπέρ 18 κατά. 139 με προφορική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ζητείτε. But it had reached the first row. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρα ψηφοφορία. 19 υπέρ, 26 κατά, παράλληλε προσπαθίε σα απορριφθήκε. Και τώρα έχουμε μία ε, επικίνδυνη ψηφοφορία για την 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 191 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά αυτό ελέγξουμε. Την 195 παρακαλώ. Πέρας. Πέρα 26 κατά απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σημείο 1 της 208 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Και αυτό έγκρινεται. Η 209 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. 210 υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 211, λέει ο πρόεδρος. Να ψηφίσουμε 211, ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται με οριακή διαφορά, λέει ο πρόεδρος. 212. 212 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή 213 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 200. 15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 217. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 υπέρ 219 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 244 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 2.59. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 2.61 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. Κατά αποχές δεκτή. 266 σε δύο κομμάτια πρώτο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 2,67 μέχρι 2,70 μπορούμε να τα ψηφίσουμε μαζί. Όχι, δεν θέλετε. 2,67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,70 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 και 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ Ναι, σωστά, έχει εκδίδει 23. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 35. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά έλεγχος για 56 Πέρας. «24-29 απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2, 3 και 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 όχι 7 δεν ψηφίσουμε έχει εκπέσει 11 mm. υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. 42 με 9 ψήφους κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Βάγκη. Και άλλοι... Ich wünsche Ihnen noch einen schönen... Καλό βράδυ σας εύχομαι. My people did not come. Yes.